Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως προβλέπει η μερίσια διάταξη, ε, έχουμε τις δηλώσεις του Συμβουλίου και τη Επιτροπής ε, για την αναστολή λειτουργίας Ελληνικού Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Θα δώσω ευθύς αμέσως τον λόγο στο Συμβούλιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Λεσκεβίσιους. Κύριε Λεσκεβίσιους. Ευχαριστώ πολύ.